Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι που παρευρίσκεστε εδώ στην αίθουσα και εκτός της αιθούσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα το όραμά μου για τις δύο βασικές πολιτικές που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό μου, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία και τις ε, διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας για αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ε, οι ειδικέ απόψεις είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση της δικής μου θέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως ειρηνευτικό σχέδιο μέσω της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Τόσο η πολιτική της διεύρυνσης όσο και η πολιτική της γειτονίας αποτελούν συνέχεια αυτού του μεγαλειώδους εγχειρήματο και στηρίζονται στις ε, θεμελιώδεις αξίες μας. Ε, θα ήθελα να ξύνω τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δύο πολιτικά πεδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει την παρουσίαση και να γίνει πιο ορατή επιτόπου, ούτως ώστε να εκπροσωπήσει τα θεμελιώδη μας ε, συμφέροντα και να λειτουργήσει σαν ε, εταίρος για την, ε, τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των γειτονικών χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξει οξύνη όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων της, θα πρέπει να έχει αυτοσυνείδηση όσον αφορά το ρόλο της ως βασικού παράγοντα στην πολιτική γειτονία και θα πρέπει να είναι αποτελεσματική στον, στην προβολή της εργασίας μας προς τα έξω. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τη διεύρυνση. Ο εκλεγμένος πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω διεύρυνση τα ερχόμενα πέντε χρόνια διότι ήρθε η ώρα να ευρωθούν τα επιτεύγματα που έχουν επιτύχει μεταξύ τους οι 28. Από ρεαλιστική άποψη, κανένα εταίρο δεν θα είναι απολύτω έτοιμο μέσα σε αυτό το διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει τέλμα στι δραστηριότητέ μα. Μάλλον το αντίθετο. Δικό μου ρόλο είναι να βοηθήσω ε, να προετοιμαστούν οι χώρε αυτέ που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, διασφαλίζοντα ότι όλα τα κριτήρια που έχουμε θέσει ε, πληρούνται. Η δική μου θητεία ως Επιτρόπου της Περιφερειακής Πολιτικής μου έδειξε την ανάγκη να προετοιμάσω νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδελεχώς για τις μελλοντικές τους ευθύνες. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία ε, κριτήρια τα οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αδιαπραγμάτευτα ή στα αγγλικά make or break για τις μελλοντικές ε, διαπραγματεύσεις ε, διεύρυνσης. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, την οικονομία και μια πλήρως λειτουργώσα δημοκρατία και βεβαίως και τις απαραίτητες δυνατότητες της διοικητικής μηχανής. Αυτά είναι καθοριστική σημασία και στις διαπραγματεύσεις μας. Το σύνθημά μου θα είναι ποιότητα και όχι ταχύτητα. Πολύ νωρί ε, στη διάρκεια τη θητεία μου θα υποβάλω προτάσει για το πώ μπορούμε να στηρίξουμε αυτέ τι προτεραιότητε για μεταρρύθμιση. Για τη δικαιοσύνη και το κράτο δικαίου θα συνεργαστώ στενά με τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον ε, Επίτροπο που θα είναι επιφορτισμένο με τα θέματα δικαιοσύνη, καταναλωτών και ισότητα των φύλων και τον Επίτροπο για τη μετανάστευση και τι εσωτερικέ υποθέσει η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, οι μεταρρυθμίσεις της, ε, του, του κλάδου της δημόσιας διοίκησης, ο ανεξάρτητος και επαγγελματικός δικαστικός κλάδος. Αυτά είναι βασικά κριτήρια για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε παραχωρήσεις. Το ίδιο και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η διακριτική μεταχείριση δεν έχει καμία θέση σε κοινωνίες που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο αδιαπραγμάτευτο ζήτημα είναι η οικονομία και οι προσπάθειές μας για ανάπτυξη και θέσει εργασία. Θα ήθελα να δω με μια νέα ματιά τα οικονομικά κριτήρια για την προσχώρηση. Α προσπαθήσουμε να αντιλήσουμε διδάγματα από την εμπειρία μα από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και να διασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια για τη διεύρυνση πραγματικά στηρίζουν του εταίρου μα, προκειμένου να επιτύχουν τα πρότυπα ε, που μια μέρα θα χρειαστούν εφόσον γίνουν μέλη και για να μπορέσουν να επιδιώξουν την ευμάρεια ήδη από τώρα. Για τις διαδοτικές μεταρρυθμίσεις προς την επιτυχία και για να είναι βιώσιμες όλες αυτές τις προσπάθειες θα πρέπει να υπάρχουν ωφέλη για τους πολίτες που να μπορούν να τα δουν και να τα κατανοήσουν. Επίση, θα φροντίσουν να υπάρξουν μεταρρυθμίσει που πρότεινα ήδη εγώ στα πλαίσια τη περιφερειακή πολιτική, ώστε να ενθαρρυνθούν οι εταίροι μα να επιδιώξουν την ανάπτυξη, εντοπίζοντα τα ε, σημεία στα οποία έχουν περισσότερες δυνατότητες από την άποψη της ανταγωνιστικότητας και με στοχοθέτηση συγκεκριμένων τομέων. Ε, για να υπάρξει στήριξη δημοσίως θα πρέπει να, δημιουργήσουμε το, ε, να στηρίξουμε το μηχανισμό για την συνδρομή πρώτης προσχώρησης μαζί με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν την κρίσιμη μάζα κέριου τομεί και να υπάρξουν πιο ορατά αποτελέσματα. Το τρίτο αδιαπραγμάτευτο στοιχείο είναι η πραγματική και ε, σε βάθο δημοκρατία. Το σώμα αυτό και τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν στη διαδικασία μεταρρύθμιση στι χώρε τη ε, διεύρυνση. Από τι δίκαιε εκλογέ, από τα πραγματικά ανεξάρτητα μέσα μαζική ενημέρωση, στην συμμετοχική και διαφανή ε, διακυβέρνηση. Ελπίζω ότι θα έχω την αμέριστη στήριξή σα. Και θα ήθελα να συνεργαστώ στενότερα και με την κοινωνία των πολιτών, ώστε αυτέ οι μεταρρυθμίσει να ριζώσουν πραγματικά. Είπε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει τελμάτωση και πράγματι, ε, υπό μία έννοια, θα ήθελα να επιταχύνουμε τις δραστηριότητές μας σε συνεργασία με τους εταίρους μας πρώτης προσχώρησης. Θα ήθελα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε την ε, περιφερειακή συνεργασία και να επιλύσουμε διμερεί ζητήματα. Οι εταίροι μας δεν μπορούν να προχωρήσουν στην ευρωπαϊκή του πορεία εάν δεν υπερβούν την κληρονομιά του παρελθόντος προηγουμένω. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιηθεί η περιοχή, ιδιαιτέρως προτείνοντας έναν εμβαθυμένο διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων υπάρχει ανάγκη για καλύτερη διασύνδεση και μεταξύ τους και με την Ένωση. Η περιοχή αυτή δεν θα πρέπει να παραμείνει μια γκρίζα περιοχή στους χάρτες των ε, οδικών, σιδηροδρομικών και ενεργειακών δικτύων. Είναι προσυφέρον όλων μας οι μεταφορές και οι ενέργειες αλλά και οι υποδομές του στα Δυτικά Βαλκάνια να ευθυγραμμιστούν με το TEN-T και το TEN-E ε ε και τα σχετικά δίκτυα. Το να έχουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους θα βοηθήσει να καταπραϊνθούν οι διασυνοριακές πολιτικές εντάσεις. Επίσης θέλω να εκμεταλλευτώ την πείρα μου ως Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής για να βεβαιωθώ ότι υπάρχουν αποτελεσματικές, σωστά ε, διαχειριζόμενες και στοχοθετημένες επενδύσεις. Θα ήθελα να υπάρξει αναζωογόνηση της συνεργασίας με την δημιουργία δικτύων στις μακροπεριοχές της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, θα εργαστώ εντατικά ώστε να πάψει η αποστράγγιση εγκεφάλων και να υπάρξει καλύτερη κυκλοφορία των υψηλών προσόντων επαγγελματιών για την επαγγελματική κινητικότητα και τα προγράμματά της. Επίσης, η Ένωση θα πρέπει να δώσει κίνητρα και για μεταρρυθμίσει στην Τουρκία. Θα ήθελα εξυγχρονισμό τη ε, ε, Τελωνιακή Ένωση, την ε, διεύρυνση των υπηρεσιών που καλύπτονται, των δημοσίων προμηθειών και των γεωργικών προϊόντων. Θα πρέπει να επιδιώξουμε από κοινού τα κοινά μα συμφέροντα, αλλά με διαπραγματεύσει προσχώρηση που θα προχωρήσουν μόνον εφόσον οι, οι τη της Τουρκίας ανεπιφύλακτα δεσμευτούν στα οικουμενικά δικαιώματα και σε μια διαρκή ατζέντα μεταρρυθμίσεων. Nation. Αξιότιμα μέλη με την ε, πολιτική γειτονία όπως ε, σχεδιάστηκε πριν από 10 χρόνια. Ποιος είχε προβλέψει την αναταραχή και την αστάθεια που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ανελαμβάνει χώρα στα νότια και τα ανατολικά της Υπήρους μας. Το να ε, αναλάβουμε αργότερο δράση στη γειτονιά μας σημαίνει ότι θα πρέπει να χτίσουμε ένα χώρο δημοκρατίας και ευημερία με μακροπρόθεσμους στόχους. Πρέπει να διαφυλάξουμε πρώτα απ' όλα την δική μας την ασφάλεια και να διαφυλάξουμε και τις οικουμενικές αξίες καθώ και τα συμφέροντά μα αμέσως. Πρώτη μου προτεραιότητα είναι να βεβαιωθούμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιληθεί η κρίση στην Ουκρανία. Συνολικό στόχο θα πρέπει να είναι μια λύση που θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τη ε, Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα και το διεθνέ δίκαιο. Θα πρέπει να στηρίξουμε το θεμελιώδες δικαίωμα της Ουκρανίας και του λαού της να ε, κάνουν τις δικές τους στρατηγικές επιλογές. Η υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας αλλά και η κύρωσή της από το σώμα σας ήταν ορόσημα. Ορόσημα που θα, φέρουν που θα ε, ενισχύσουν τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας αλλά θα προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ευημερία και στην Ευρωπαϊκή Πύρο συνολικά. Η συμφωνία αυτή είναι ένα απαραίτητο πλαίσιο για τις δεσμεύσεις μας στα ανατολικά και τα νότια. Ωστόσο θα πρέπει να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ο πρόεδρος Γιούνκερ μου ζήτησε να προτείνω συστάσεις κατά το πρώτο έτος της θητείας μου. Θα ήθελα να υπάρξουν ευρύτατες διαβουλεύσεις γι' αυτό με τη δική σας συμμετοχή, αλλά ορισμένα στοιχεία είναι ήδη πολύ σαφή. Πρώτον, Ανέκαθεν λέγαμε ότι η πολιτική αυτή, η πολιτική της γειτονίας θα πρέπει να ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση για κάθε χώρα. Αυτό τώρα θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Δεύτερον, η πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι πιο διαλλακτική και ευέλικτη και να δίνει άμεσες απαντήσεις όταν μας χρειάζονται οι εταίροι μας. Τρίτον, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τη συνεργασία μας σε όλα τα βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, του εμπορίου και της μετανάστευση. Τέταρτον, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανάληψη ευθύνη από κοινού στι σχέσει μα με του γειτονέ μα. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών υπό την ευρύτερη έννοια συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων. Επιτρέψτε μου να πω και το εξή. Όταν οι εταίροι μα με καλύτερη διακυβέρνηση και μεταρρυθμίσει δίνουν καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατήσει τι υποσχέσει τη. Όταν οι εταίροι μα δεν επιτυγχάνουν τα κατάλληλα αποτελέσματα, θα πρέπει να έχουμε μια σαφή στρατηγική ώστε να επιδιώξουμε τα δικά μας συμφέροντα και να διατηρήσουμε την επιρροή μας παραμένοντας πιστοί στις αξίες μας και στις αρχές μας. Προς Ανατολάς, η ανατολική γειτονία και η πολιτική της ε, προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο που θα πρέπει να προσαρμόζεται στα γεγονότα. Ε, θα ήθελα να βεβαιωθώ ότι η Ουκρανία, η Γεωργία και η Μολδαβία θα λάβουν όλη τη στήριξη που χρειάζονται για να κάνουν τις δικές τους δημοκρατικές επιλογές και να αναλάβουν τις απαραίτητες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Η ομάδα στήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ουκρανία θα καθορίσει έναν ε, βασικό ρόλο για το έργο μα εκεί, μαζί με την ανοικοδόμηση τη Ανατολική Ουκρανία. Θα ήθελε να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν και θα ήθελε επίση να ε, ενταθεί η πολιτική συνεργασία για την ε, σχέση μα με την ε, Θα στηρίξω τι προσπάθειε τη Φεντερίκα Μογκερίνη, ώστε ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχυθεί και να συμβάλλουμε στην επίλυση των παγωμένων συγκρούσεων στην ανατολική γειτονιά μα. Μαζί με την ε, ε, είπα το εκπρόσωπο θα ήθελα να προωθήσουμε το διάλογο και με τη Ρωσία. Δεν θα πρέπει να υποτιμά την ε, απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει πιστή στις αξίες της η Ρωσία και θα πρέπει να κατανοήσει η πολιτική, ότι η πολιτική γειτονία μας και οι εταιρικέ σχέσεις προς Ανατολάς δεν θα υλοποιηθούν εις βάρος της Ρωσίας. Και τώρα προς τον Νότο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ως προς την αρχή της, διαφοριο... της διαφοροποίησης. Και έχω κατά νου εταίρους που έχουν φέρει εις πέρας διαρκείς μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένα ε, και μακρο... με βιώσιμα αποτελέσματα, ιδίως στην Τινησία και το Μαρόκο. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι εταίροι αυτοί μπορούν να περάσουν σε δημοκρατικό διάλογο, να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρξει ειρήνη και ευημερία στην περιοχή. Στη Συρία έχουμε τεράστια πολιτικά και ανθρωπιστικά προβλήματα μια τεράστια κρίση. Δεν θα πρέπει να επισκιαστεί το πρόβλημα αυτό από άλλε αναταραχέ σε άλλα μέρη τη γειτονιά μα. Θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειε για την ε, εξέβρεση πολιτική λύση και να πάψει ο πόνο αυτού του λαού των κοινοτήτων σε αυτή την περιοχή αλλά και στην Ιορδανία και το Λίβανο. Στην Αίγυπτο είναι περίπλοκη πολιτική κατάσταση και το πολιτικό τοπίο και πολύ δύσκολε οικονομικέ συνθήκε που ε, δείχνουν ότι χρειάζεται κρίσιμη και επικοδομητική ανάλυση ε, δεσμεύσεων και για την Λιβύη θα πρέπει να εμποδίσουμε να επέλθει το χάος στη χώρα αυτή, να στηρίξουμε τις αρχές και να υπάρξει πολιτικός διάλογος για μια μετάβαση προς μια διαρκή σταθερότητα. Επίσης η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαδικασία ειρήνευσης στην, Ανατολική, στην Μέση Ανατολή θα πρέπει να συνεχιστεί σε συνεργασία με την κυρία Μογκερίνη με όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αξιότιμα μέλη. Δύο λόγια μόνο για, την, για, τον ε, ευρωπαϊκό χώρο, για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τον ε, Χώρο Ελεύθερου Εμπορίου. Μαζί με την ΕΠΑΤΟ εκπρόσωπο θα συνεργαστούμε με τους βασικότερους εταίρους μας ώστε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στην εσωτερική αγορά και να γίνονται σεβαστές οι τέσσερις βασικές ελευθερίες μας, χωρίς ιδιαίτερες επιλογές. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινωνία της αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις σε μια εποχή στην οποία είναι περιορισμένα τα οικονομικά μας μέσα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευθύνη της εστιάζοντας περισσότερο στην πολιτική γειτονίας και διεύρυνσης. Θα ήθελα λοιπόν να συνεργαστώ στενά με την Επιτροπή σας για να διασφαλίσουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να δρά προληπτικά και στοχευμένα για το καλό των πολιτών μας. θα αναλάβω καθήκοντα με ενθουσιασμό αλλά και ρεαλισμό. Ας συνεργαστούμε με αποφασιστικότητα και ρεαλισμό για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους ε, γείτονές μας ε, πάντα προς τα ε, ευρωπαϊκά μας συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ.